μός σε μια επιτροπή θα καταγραφεί στα πρακτικά. Αν δεν υπάρχει καμία άλλη παρατήρηση, ο οδηγισμός αυτός θεωρείται εγκεκριμένος. Ευχαριστώ πολύ.